Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πάρτε τις θέσεις σας. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Προχωρούμε στις ψηφοφορίες. Πριν από αυτό έχει ζητήσει το λόγο για point of order ο κύριος Αχματ Μπασίρ. Παρακαλώ κύριε Μπασίρ, έχετε το λόγο. Κύριε συνάδελφοι, παρακαλώ να ακούσουμε τον κύριο Αχματ Μπασίρ.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 it's a, chair. Αξιότιμε πρόεδρε. Χθες στο Sky News είδαμε είδε ο κόσμος πόσο υποφέρουν οι Ραχίγκα. Εγώ το είδα από πρώτη ματιά, πρώτο χέρι, όταν συνάντησα τους επιβιώσαντες της γενοκτονίας των Μπαγκλαντές. Στο Μιανμάρ γεννούνται μωρά στην παραλία. Οι τυχεροί θα πάνε σε βαπόρι, σε βάρκα και θα πάνε στον Μπαγκλαντές. Οι υπόλοιποι θα μείνουν να πεθάνουν. Η Βρετανίδα Πρωθυπουργό υποσχέθηκε να αντιμετωπίσει αυτή την απάνθρωπη καταστροφή των Ραχίνγκα. Απευθύνω έκκληση μόνο ο πρόεδρος να δώσει άδεια για έκτακτη συζήτηση για να εξετάσουμε την κατάσταση των Ραχίνγκα σύμφωνα με το άρθρο 153 παράγραφος 4 διότι μετά από μακροσκελή συζητήσει με τον ΟΗΕ, το Μιανμάρ, τον Μπαγκλαντές και τον Ομένο Βασίλειο, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει τώρα να συγκαλέσει μια διακυβερνητική σύνοδο κορυφή για να τεθεί τέρμα σε αυτή τη γενοκτονία. Για λόγους, της για λόγους ανθρωπισμού και για την ανθρωπότητα συγγυηθεί το Κοινοβούλιο σε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ. Κύριε Μπασίρα, άκουσα με προσοχή την πρότασή σας και τους λόγους που την στηρίζουν. Αυτό που δεσμεύομαι είναι να διαβιβάσω αμέσως στον Πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου την πρότασή σας. Προχωρούμε τι ψηφοφορίες. Έκθεση Διώτη, κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας.